Bene, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Λοιπόν, καλό απόγευμα σε όλες και όλους, λέει ο Πρόεδρος. Να καλωσορίσω στο δεύτερο αυτό τμήμα της εκδήλωσης Αχάροφ αφιερωμένο στις Ομικρών, που λειτουργούν στην Μεσόγειο σώζοντας ανθρώπινες ζωές η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με τις ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές ε, δικαιωμάτων του ανθρώπου, εσωτερικών υποθέσεων και δικαιοσύνης. Στα αριστερά μου ο συνάδελφος Κλοντ Μωράης, πρόεδρος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Μαζί, από κοινού, θα προεδρεύσουμε στη σημερινή συνάντηση. το πέρασμα αυτό της ε, Μεσογείου έχει καταστεί πολύ επικίνδυνο εγχείρημα για έναν αριθμό μεταναστών που επιχειρούν να έρθουν στην Ευρώπη ψάχνοντας καλύτερες συνθήκες ζωής και μεγάλο μέρος τους ανθίσταται σε, αυτήν την, σε αυτόν τον κίνδυνο για ένα ταξίδι που γίνεται υπό πολύ δύσκολες συνθήκες και υπό τη διοργάνωση λαθρεμπόρων που δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Οι μη καπόμικρον λοιπόν σώζουν πολλούς από τους ανθρώπους αυτούς από τη θάλασσα, πάρα πολλούς τα τελευταία χρόνια. Η Υποεπιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προ δύο εβδομάδων επισκέφθηκε την ε, Ρώμη για να ελέγξει ποια είναι η κατάσταση των προσφύγων και μεταναστών. Στην αποστολή αυτή είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε κάποιες μικρά από που είναι σήμερα οι εκπρόσωποι τους εδώ μαζί μας εξάλλου και που μας ε, έδωσαν ένα, μια συνολική εικόνα των συνθήκων υπό τις οποίες ε, ε, λειτουργούν. Επίσης είχαμε τρομακτικές μαρτυρίες από μετανάστες και πρόσφυγες από άνω των 20 χωρών, σε όλες αυτές τις επαφές και συναντήσεις υπογραμμίστηκε, σημειώθηκε η καταστροφική κατάσταση ε, που επικρατεί στη Λιβύη. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα μας φάνηκε σημαντικό να ακούσουμε ζωντανά τις μαρτυρίες αυτές και στην, στο πρώτο μέρος της συνάντησης αυτής ε, θα μας διηγηθεί την ιστορία τη δική του ο Φίλιμον Μπράτο από την Ερυθρέα και το επικίνδυνο ταξίδι, διαδρομή που έκανε στη Μεσόγειο. Θα ακούσουμε και την μαρτυρία της Κάτριν Σμιτ, μέρος του πληρώματος Γιουβέντα που συμμετείχε στις ε, επιχειρήσεις διάσωσης. Χωρίς άλλη καθυστέρηση θα δίνω αμέσως το λόγο στον ε, Φίλιμον Μεμπράτομ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ που με επιτρέπετε να ήρθω ενώπιον σας και να μπορέσω να σας πω την ιστορία μου. Την ιστορία μου. Είμαι από την Ερυθρέα. Από την πατρίδα μου και τους ανθρώπους της, την φύση, την μουσική, λέγω μερατόμ. Όλα αυτά μου λείπουν εδώ στην Γερμανία. Παρ' όλα αυτά αναγκάστηκα να καταλήψω την αγαπημένη μου πατρίδα διότι ήθελα να ζήσω ελεύθερος. Ενώ εκεί υπάρχει και κίνδυνος για τους νέους ανθρώπους διότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν σημαίνουν τίποτε και δεν υπάρχει ελευθερία έκφρασης. Καμιά ελευθερία δεν υπάρχει στη χώρα αυτή. Όσο θυμούμε τον εαυτό μου, έχω ζήσει μόνο δυστυχία και βία. Οι στρατιώτες έρχονται και παίρνουν τους ανθρώπους με το ζόρι στο στρατό, ακόμα και μικρά παιδιά. Ποιος ξέρει τι συμβαίνει με, με τους ανθρώπους αυτούς πρόκειται για δικτατορία και ο δικτάτορα κάνει ό,τι θέλει, καταπιέζει τον λαό του. Εγώ έκανα μια εκπαίδευση εκεί ε, ως ε, φωτογράφος, κάμεραμαν και ήθελα να γίνω δημοσιογράφος για να δείξω στον κόσμο την αλήθεια. Αλλά μέσα στην δικτατορία αυτή δεν βρήκα καμιά ελπίδα να εργαστώ ως δημοσιογράφος. Θα σήμαινε διαρκή κίνδυνο, ίσως και θάνατο. Η φυγή μου με οδήγησε μέσω Αιθιοπίας, Σουδάν και την έρημο. Κόντεψα να πεθάνω από την δίψα. Θυμόμουν την αγαπημένη μου μητέρα, η οποία όταν ε, πεινούσα ή διψούσα με φρόντιζε. Τώρα περνώ μέσα από την έρημο χωρίς τροφή, χωρίς νερό. Στην έρημο πεθαίνουν πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν θάβονται καν. Παραμένουν εκεί, στην άμμο, παντού βλέπει κανείς ε, μουμιοποιημένα πτώματα. Αυτό μου έκοψε τη λαγιά. Για να φτάσω χρειάστηκε να πουλήσω τη ζωή μου. Με πουλήσανε σαν να είμαι κανένα λαχανικό. Είμαι άνθρωπος όμως. Πέρασα από διάφορα στρατόπεδα και τα πράγματα που έζησα εκεί για μένα ήταν η κόλαση. Χτυπούν τους ανθρώπους καθημερινά, τους πυροβολούν. Σε ένα από τα στρατόπεδα αυτά ζουν 4.000 άνθρωποι. Πολλοί από αυτούς θα πεθάνω από πείνα και δίψα. Όταν δεν έχουμε άλλη επιλογή, σπάμε την πόρτα για να βγούμε έξω. Καμιά φορά βάζουν και φωτιά οι φρουροί στα, στα στρατόπεδα. Δηλαδή εμπρισμούς. καταφέρουν να φτάσουν στην παραλία και έρχονται τότε οι διακινητές μας αναγκάζουν να περάσουμε από το νερό. Το μαύρο νερό με φοβίζει, είναι νύχτα. Ποτέ δεν έχω βρεθεί στη θάλασσα, δεν ξέρω να κολυμπώ. Μας βάζουν να σταθούμε σε μια σειρά, εγώ είμαι από τους πρώτους. Επειδή όμως έχω τόσο μεγάλο φόβο, με βάζουν πίσω. Δεν είμαι βέβαιος αν θα μπορέσω να επιζήσω. Μας βάζουν πρώτα σε ένα φουσκωτό σκάφος και μας φέρνουν σε αυτό σε ένα ξύλινο, το οποίο είναι υπερπλήρες αισθάνομαι αβοήθητος. Οι διακινητές με αναγκάζουν να μπω στο αμπάρι. Εκεί είναι πραγματική κόλαση. Δεν έχω αέρα, δεν παίρνω αέρα. Προσπαθώ να κρυφτώ ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους. Έχω πληρώσει τόσα λεφτά. Γιατί είμαι υποχρεωμένο τώρα να πεθάνω μέσα σε αυτό το αμπάρι. Εν τέλει βρίσκω κάποια θεσούλα που μπορώ να καθίσω. Η θάλασσα είναι ταραγμένη. Τα κύματα κουνούν το σκάφος. Πολλοί κάνουν εμετό. Άλλοι πνίγονται από τους εμετούς του. Εγώ φοβούμαι πολύ, αλλά πρέπει να επιζήσω. Κάποια στιγμή βγαίνει ο ήλιος. Μετά από πολλές ώρες στη θάλασσα. Εγώ έχω χάσει κάθε ελπίδα και θεωρώ ότι θα πεθάνουμε. Τα σκοτεινά νερά μου προκαλούν πανικό. Μέσα στο σκάφος είναι και οι γυναίκες. Μια γυναίκα με τέσσερα παιδιά. Άνθρωποι τραυματίες. Εγώ ανησυχώ πολύ για τα τέσσερα παιδιά. Εγώ είμαι μόνος από την οικογένειά μου στο σκάφος αυτό. Το απόγευμα μας διασώζει πλοίο του Ιταλικού Ναυτικού. Είμαι πια πολύ χαρούμενος. Θεωρώ ότι σώθηκα από αυτά τα βαθιά ε, σκοτεινά νερά. Αυτά φθινόπωρο του 2014. Σήμερα θα ήταν αλλιώ τα πράγματα. Να περάσει κανείς στη Μεσόγειο με ένα φουσκωτό σκάφος ή με ένα χαλασμένο ξύλινο σκάφος. Αυτό θα σήμαινε για μένα ότι χάνω τη ζωή μου και τη δυστυχία στην οικογένειά μου. Δεν υπάρχει η ευκαιρία να περάσω με ένα σωστό σκάφο στην Ευρώπη ή με ένα αεροπλάνο. Εντελώ αβοήθητο. Τι μπορώ να κάνω για να φτάσω σε ασφάλεια. Ο κάθε άνθρωπο μια ζωή έχει, όπω και εγώ. Κάθε άνθρωπο θέλει να ζήσει τη ζωή του σε ελευθερία. Όπω ένα λευκό περιστέρι θέλει να πετάξει όπου μπορεί. Εγώ διακινδύνευσα τη ζωή μου για να έρθω στην Ευρώπη παρόλο που δεν με δέχτηκαν στη Γερμανία. Είναι πολύ στενά ε, περιορισμένη η ζωή μου στη Γερμανία. Από το 2014 ζω στη Γερμανία χωρίς διαβατήριο. Δεν ξέρω ακόμη πόσο θα μου επιτρέψουν να ζήσω στη Γερμανία και πότε θα με απελάσουν. Και πού να πάω. Τι σας έκανα. Στο κάτω είμαι και εγώ, στο κάτω είμαι και εγώ άνθρωπος όπως εσείς. Κάθε μέρα πεθαίνουν τόσοι χιλιάδες άνθρωποι στη Μεσόγειο. Όλοι εσείς εδώ στην Ευρώπη περνάτε καλά. Η Ευρώπη έχει κλειδιά στα χέρια της για να ανταλλάξει όλα αυτά τα πράγματα και να σταματήσει το θανατικό αυτό. Γιατί δεν το κάνετε. Γιατί αφήνει τους ανθρώπους να πεθαίνουν. Μέχρι πότε θα πρέπει να πεθαίνουμε στην, πάνω στην φυγή και να πεθαίνουμε από τη δίψα στην έρημο ή να πνιγόμαστε στη Μεσόγειο. Μέχρι πότε θα πρέπει να περιμένουμε για να μας αναγνωρίσουν ως ανθρώπους. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη μαρτυρία σας. Η Κάτριν Σμίτ έχει το λόγο τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ τον να καταρχά, που ήρθε σήμερα εδώ και μας μίλησε και ευχαριστώ και για την πρόσκλησή σας ε, να μιλήσω ενώπιον σας σήμερα. Μου ζητήθηκε να μιλήσω για τις εμπειρίες μου ως μέλος του πληρώματος του Ιουβέντα στην διάσωση στη θάλασσα και ως μάρτυρας ε, της, ε, των εξελίξεων στην πόρτα μας. Ούτε ναυτικός είμαι, ούτε έχω ασχοληθεί ε, με, είχα πιστέψει ότι θα σχολιόμουν ποτέ με το θέμα της διάσωσης στη θάλασσα. Ωστόσο, αποφάσισα να ασχοληθώ με το θέμα της διάσωσης στη θάλασσα γιατί πεθαίνει ο κόσμος. Ίσως να χρειαστεί να δικαστώ μαζί με άλλα εννέα μέλη του πληρώματος του Ιουβέντα γιατί δώσαμε στους ανθρώπους αυτούς το βασικό δικαίωμά τους που δεν τους έδωσε μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, το δικαίωμα στη ζωή, προστατεύοντας την ανθρώπινη ζωή και τις αξίες της Ευρώπης τώρα ορίζεται ως υποστήριξη της παράνομης μετανάστευσης και ε, υφίσταται τον κίνδυνο να μας, φέσει, να μας φυλακίσει για 20 χρόνια. Ανθρώπους οι οποίοι πνίγονται ε, κάτι που βιώνουμε σε καθημερινή βάση και είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό. Κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε χωρίς να σκεφτούμε δύο φορές. Σώσαμε σώζοντας αυτούς που πρέπει να σώζουμε, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό δεν μπορεί ποτέ να τεθεί υπό την αίρεση πολιτικών συζητήσεων, ωστόσο μπορεί να δικαστούμε επειδή σώσαμε 14.000 ανθρώπους στη θάλασσα. Ωστόσο, το θέμα δεν είναι ε, η ποινικοποίηση της δράσης αυτής. Αυτό που είναι πιο σημαντικό και θέλω να πω σήμερα είναι να μιλήσω στο όνομα των λιγότερων προνομιούχων που συνεχίζουν να πεθαίνουν κάθε μέρα προσπαθώντας να φτάσουν με ασφάλεια στις ευρωπαϊκές ακτές. Είμαι μέλος μιας γενιάς που μεγαλώσε ρωτώντα τους παππούδες μας τι κάνατε κατά της βίας στον πόλεμο. Είμαι τώρα ανήκω σε αυτήν την γενιά που θα πρέπει να απαντήσει τώρα στα δικά μου εγγόνια όταν με ρωτήσουν τι κάνατε την περίοδο εκείνη. Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις και τα κράτη-μέλη της Ένωσης ήταν αυτά που όχι μόνο απομάκρυναν τη Γιουβέντα από εκεί που ήταν πιο αποτελεσματική, αλλά ξεκίνησαν ποινικέ διαδικασίες, άσκησαν, ασκήθηκε ποινική αγωγή, ποινική δίωξη εις βάρος μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πίεσε την Ιταλία, τις Ιταλικές αρχές να συμφωνήσουν με αυτούς που, από τους οποίους προστατεύουμε τους ανθρώπους. Την ακτοφυλακή της Λιβύης που στην πραγματικότητα είναι διακινητές που χρηματοδοτούνται για να πάρουν πίσω τους ε, μετανάστες και πρόσφυγες και να αντιμετωπίσουν στην, την βία, τη, τα βασανιστήρια και το θάνατο στη Λιβύη. Η Ευρώπη είναι υπεύθυνη για εγκρήματα κατά της ε, ανθρωπότητας. Εμείς ε, επιτρέπουμε στους, ε, στην ακτοφυλακή της Λιβύης να δράσει το όνομα της Ευρώπης, να πυροβολούν ανθρώπους στη θάλασσα, στο νερό, να σκοτώνουν εσκεμένα άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη. Το χέρι της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραβιάζει συνεχώς τους κανονισμούς που ε, αποτέλεσαν την βασική, το βασικό πολιτικό ε, επίτευγμα της εποχής μας, την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η Ιουβέντα βλέπει τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου που ασκούν η Λίβοι κάτω από την αιγίδα ενός ευρωπαϊκού προγράμματος. Οι νέες μας φυλακές αποτελούν, ε, οι νέες μας πιέσεις πρέπει να αγνοηθούν. Η ιστορία του πληρώματος, η ιστορία της Γιουβέντα είναι και δική μου ε, ιστορία. Θυμίζει ένα κακό αστυνομικό μυθιστόρημα. Το Μάιο του 2017, το Κέντρο Συντονισμού Διάσωσης της Ιταλίας αντιμετώπισε μία από τις πιο ε, δύσκολες ε, δραστηριότητες της, την υποχρέωσή της να απομακρύνει το Γιουβέντα από την περιοχή διάσωσης στην, ε, μας οδήγησαν, μας, μας ε, ε, υποχρέωσαν να μην βοηθήσουμε όσους ε, πνίγονταν ή βρίσκονταν σε κίνδυνο εκείνη τη στιγμή. Η Γιουβέντα χρειάστηκε να ακολουθήσει τις εντολές των Ιταλικών αρχών και μετά από 48 ώρες, μετά από 48 ώρες στις 2 και 40 το πρωί κοντά στη Λαμπεντούζα στην γέφυρα του πλοίου διαπιστώθηκε ένας, ότι βρέθηκε, υπήρχε ένας κοριός των Ιταλικών αρχών πάνω στη γέφυρα του πλοίου. Εγώ και άλλα δύο μέλη του πληρώματος χρησιμοποιήσαμε αυτή τη διαδικασία για να βοηθήσουμε άλλες, ε, άλλα πλοία ΜΚΟ για την προσπάθεια διάσωσης. 21 σκάφη με χιλιάδες μετανάστες εμφανίστηκαν όταν ξημέρωσε. Πραγματικά εκείνη τη στιγμή χρειαζόταν κάθε άνθρωπος και κάθε σωσίβιο θα μπορούσε να είχε ε, χρησιμοποιηθεί. Την ίδια στιγμή οι Ιταλικές αρχές είχαν κρατήσει στη βία στο λιμάνι της Λαμπεντούζα σκάφη που είχαν εκατοντάδε σωσίβια. Μετά από αυτέ τι τέσσερι ημέρε, η χειρότερη στιγμή ήταν όταν διαπιστώσαμε πω είχαμε χάσει πέντε σκάφη με πάνω από 800 άτομα μετά από αυτή την ε, τρικυμία, εκείνη τη νύχτα. 600 άτομα είχαν χαθεί στη θάλασσα χωρί ίχνους. Μπήκαν απλά στι στατιστικέ των ε, χαμένων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. μαζί με τους αγνοούμενους χάθηκαν και οι αξίες της Ευρώπης. Έτσι έμαθα να καταλαβαίνω τα άθλια αίτια της συστηματικής άρνησης δικαιωμάτων και βοήθεια σε άτομα που χάνονται είτε στη θάλασσα είτε στα κέντρα κράτησης της, Ιβύλης, της Λιβύης. Η στρατηγική αυτή είναι μια σκεμμένη στρατηγική που μετατρέπει τη Μεσόγειο σε, στην πιο ε, φωνική θάλασσα του κόσμου. Τρεις μήνες μετά τις ε, προσπάθειες που έκαναν οι Ιταλικές αρχές να βάλουν κοριού στο σκάφος μας, το Ιουβέντα, ε, υποχρεώθηκε να επανέλθει στο λιμάνι της Λαμπεδούζας, όπου της έγινε έρευνα. Α, αντιμετωπιστήκαμε με προληπτικά μέτρα και βάση της ε, νομοθεσίας κατά, για την καταπολέμηση της μαφίας λίγες μέρες αφότου είχαμε διασώσει 3.500 άτομα μετά από εντολή και με συνεργασία με την Ιταλική Ακτοφυλακή. Τότε ήμουν επικεφαλής αποστολής στη Γιουβέντα. Το πλοίο μας είχε ε, ερευνηθεί για όπλα από 15 αστυνομικούς. Τα προσωπικά μας ήδη κατασχέθηκαν, ακόμα και σήμερα δεν έχουν δοθεί. Ε, μετά από την έρευνα φαινόταν, το, το πλοίο φαινόταν σαν να είχε πληγή από τη τυφώνα. Τα μέτρα αυτά, το πιστεύω ακόμα περισσότερο τώρα όπως και τότε, ότι ως, ο μόνος στόχο είχαν να μας εμποδίσουν να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Η, επί, η εγώ αντιμετωπίστηκα ως εγκληματίες γιατί προσπαθούσαν να σώσουν ανθρώπους. Ο, απλώς γιατί παρενέβην όταν οι ίδιες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που υποστηρίζουν θεωρητικά τις ευρωπαϊκές αξίες τις καταπατούν και αφήνουν τον κόσμο να πεθάνει. Η κοινωνία των πολιτών είναι αυτή μόνο που μπορεί να προστατεύσει τους ανθρώπους αυτούς. Δεν μπορούν να εμποδίζεται και να υποτιμάται η δουλειά των ΜΚΟ. Τους τελευταίους 20 μήνες το Ιουβέντα έχει, ε, είναι δεσμευμένο στο λιμάνι του Τράμπανη και δεν μπορεί να σαλπάρει με εντολή των Ιταλικών αρχών. Προσφέροντας ε, η, η προσπάθειά μας να βοηθήσουμε απλά τους άλλους υπόκειται σε ποινική δίωξη. Εγώ έχω όμως τη δική μου καταγγελία να κάνω, ότι αυτή τη στιγμή κατηγορώ όλους αυτούς οι οποίοι ε, επικαλούνται την ευρωπαϊκή ε, νομοθεσία, ότι δεν σέβονται την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ότι στέλνουν τους ανθρώπους στο θάνατο στη θάλασσα ή στα ε, στρατόπεδα θανάτου της Λιβύης, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο. Αυτό που διακυβεύεται στην έρευνα αυτή ξεπερνά τις προσωπικές την προσωπική ελευθερία των, ε, του πληρώματος του Γιουβέντα. Η προσπάθεια διάσωσης ανθρώπων θεωρείται ως πολιτικό εργαλείο και η προσπάθεια των δικαιωμάτων του ανθρώπου θεωρείται ως παραβίαση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Αυτό σημαίνει ότι τίθεται σε κίνδυνο η τίθεται σε κίνδυνο όλες μας οι αξίες. Αυτό που αυτό, που κατηγορείται, αυτό για το οποίο κατηγορούμαστε είναι γιατί προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε αυτούς που να διασώ, και διασώσαμε αυτούς που κινδύνευαν να ε, πεθάνουν. Και αυτό από αυτούς οι οποίοι εμποδίζουν την διάσωση αυτών των ανθρώπων. Ένας τέτοιος κόσμος δεν είναι ένας κόσμος στον οποίο θα ήθελα να ζω. Δεν φοβόμαστε ούτε από τις ε, καμπάνιες ε, ε, που μας καθιστούν λιγότερο δημοφιλείς, ούτε με καμπάνια παραπληροφόρησης. Ξέρουμε ότι η κατάσταση μπορεί να γίνει πολύ πιο δύσκολη. Κάνω έκκληση στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην κοινωνία των πολιτών. Μην αγνοείτε αυτή την δυσάρεστη πραγματικότητα. Αναγνωρίστε το δικαίωμα του καθενός, αναγνωρίστε τις ευθύνες όλων για τους μαζικούς θανάτους στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και κάντε κάτι για να σταματήσουν οι θάνατοι αυτοί, ώστε να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη στην οποία οι άνθρωποι που έρχονται αναζητώντας αξιοπρέπεια και ε, ζωή θα μπορέσουν να ζήσουν ως ελεύθεροι άνδρες και γυναίκες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κάτριν για την παρέμβασή σου. Οι βουλευτές Κάποιες παρατηρήσεις, σχόλια. Η αναγκόμες. Thank you so much for... Ευχαριστώ πολύ για τις μαρτυρίες σας και τους δύο. Και ε, πραγματικά ήταν συγκλονιστικές. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αισθάνομαι τροπή που έτσι είναι η κατάσταση στην Ευρώπη αυτές τις μέρες. Και αποτείω και φόρο τιμής σε ανθρώπους όπως εσείς κυρία Σμιτ που παρόλε τις δυσκολίες, τις παρενοχλήσεις επιμένετε να αγωνίζεστε για να διασώζετε ζωές και έτσι και την αξιοπιστία μας. Αισθάνομαι αγανάκτηση που η mainstream πολιτική και οι κυβερνήσεις στην ουσία μόνο λόγια λένε για την κρίση του μεταναστευτικού, ενώ στην πραγματικότητα είναι κρίση της πολιτικής και κρίση των αξιών τους, που αγνοούν τις βασικές αξίες του ευρωπαϊκού εγχείρηματος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. δυσκολεύομαι να καταλάβω πώς τους τραβάει από τη μύτη αυτή η ξενοφοβική άκρα δεξιά, αυτές, αυτά τα ψέματα που λέει. Γιατί είμαστε σε μια Ήπειρο όπου χρειαζόμαστε τη μετανάστευση, τους χρειαζόμαστε τους μετανάστες, ακόμα και αν είναι μόνο για να κρατήσουμε στα πόδια του ή στα πόδια τους τα ε, συστήματα κοινωνική ασφάλεια για να αντιμετωπιστεί η γύρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Χρειαζόμαστε μετανάστες όπω ο Μερατόμ που έχει το θάρρο να φύγει για να προσπαθήσει να ζήσει σε ελευθερία και αξιοπρέπεια. Άνθρωπο είναι όπω και εγώ. Και θέλει να ζήσει σε συνθήκε ελευθερία και αξιοπρέπεια όπω και εγώ. Και γι' αυτό εγώ ζω στην Ευρώπη. Και έχει δίκιο που λέει ότι η Ευρώπη έχει τεράστια ευθύνη και θα μπορούσε και θα πρέπει να αλλάξει τα πράγματα. Θα ήθελα μόνο με την ευκαιρία να ζητήσω και από εσά και τους δυο σας και από τους δυο σας και νομίζω ότι είπατε και εσείς κυρία Σμίτ όλη αυτή η ψευδολογία που συνεχίζει και ακόμα και εδώ μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ισχυρίζεται ότι υπάρχει ένα τι να πω, μια λιβική ακτοφυλακή, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για πολιτοφυλακές, για μιλήσια, για ένοπλες ομάδες που εμείς τους αποκαλούμε λιβική ακτοφυλακή. Αλλά αυτοί είναι οργανωμένες ομάδες οι οποίες αυτές μάλιστα οργανώνουν τις διακινήσεις των μεταναστών και εκμεταλλεύονται με τον χείριστο τρόπο ανάγκες όπως του κ. Μερατόμ ή των άλλων που θέλουν να ζήσουν σε ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σουσνιέλτς. Ε, το Ευχαριστώ, πρόεδρε. Αυτά που ακούμε εδώ είναι απολύτως ε, δημαγωγικά. Ακούμε ιστορίες που είναι συγκινητικές ε, και υποτίθεται ότι μας πείθουν μάλλον αυτό προσπαθούν να κάνουν, αλλά εδώ ακούμε για ανθρώπους που δολοφονούνται, άνθρωποι που προσπαθούν να ζήσουν ειρηνικά σε ελληνικά νησιά και τους επιτίθενται κτλ. Έχουμε παραδείγματα τέτοια ιδιαίτερα επίσης συγκινητικά, αλλά ε, δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο ρόλος του νομοθέτη. Ο ρόλος του νομοθέτη είναι να διατηρεί την ψυχραιμία του, να κοιτάζει τα πράγματα όσο αναλυτικότερα μπορεί και να βλέπει τι κάνουν οργανώσεις όπως αυτή που χειρίζεται το Ιουβέντα. Εάν το μήνυμα που διαβιβάζουμε στους ανθρώπους αυτούς είναι ότι περιπολούμε τις ακτές, τότε αποθαρρύνουμε τους λαθρεμπόρους ενδεχομένως. πάντοτε θα έχουμε ε, μια επιθυμία να προσέρχονται άνθρωποι από πιο φτωχές χώρες, από εμπόλεμες ζώνες, σε μια καλύτερη κοινωνική κατάσταση. Και δεν μιλούμε για χώρες μόνο όπως η Λιβύη. Υπάρχουν ε, ροές που προέρχονται από το ίμιση της Αφρικανικής Υπήρου. Δεν είναι μόνο δηλαδή άνθρωποι που διαφεύγουν, προσπαθούν να σωθούν δηλαδή από πολεμικές συγκρούσεις. Η κυρία Γκόμες, εφόσον μας λέει ότι χρειαζόμαστε εκατομμύρια μετανάστες, ίσως ε, να μην τους χρειαζόμασταν αν δεν δολοφονούσαμε τα ίδια τα δικά μας τα αγέννητα παιδιά. σε εκείνους δηλαδή που διενεργούν ε, αμβλώσεις παράνομες διακόπτη ο πρόεδρος, συνεχίζει ο μιλητής. εσείς στερείτε ε, ε, τα παιδιά αυτά από το δικαίωμα στη ζωή, στερείτε ε, το μέλλον από την Ευρώπη. Αποθαρρύνουμε τους ανθρώπους από το να δουλεύουν και από το να φροντίζουν τα δικά τους παιδιά. Και δεν τους δίνουμε τα μέσα, μάλιστα. νομίζω ότι πρέπει να έχετε αξιοπρέπεια, λέει ο Πρόεδρος. Δεν είναι ηρωνικά αυτά που λέω, είναι επιχειρήματα λέει ο Λοιπόν, η κυρία ε, Ρούιθ, ε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ δεν είχα την πρόθεση να ζητήσω το λόγο γιατί έφτασα αργά και δεν είχα την ευκαιρία να ακούσω όλη την ε, παρουσίαση, την εισήγηση. Αλλά αφού μας λένε εδώ συνάδελφοι ότι θέλουν επιχειρήματα, να τους δώσουμε. Πρώτον, δεν ξέρω αν είστε ειδικό στα θέματα της τρομοκρατία. εγώ είμαι. Κατά και πολλών ετών έχω διάφορα παράσημα μετάλλια, συνταγματικό μεταξύ άλλων της χώρας μου, για την προσπάθειά μου, για τον αγώνα μου, για την προστασία των θυμάτων της τρομοκρατίας. Κάτι ξέρω για την τρομοκρατία. Και εγώ μπορώ να σας πω ότι αυτά που είπατε εσείς είναι απολύτω αβάσιμα. Έχουμε πάρα πολύ λίγες περιπτώσεις ανθρώπων που χρησιμοποίησαν δίκτυα παράνομης μετανάστευση προκειμένου να διαπράξουν εγκλήματα. Αυτά που είπατε εσεί είναι απολύτω ψευδή. Αυτό είναι το πρώτο. Και εγώ ξαναλέω, είμαι ειδική στα θέματα ε, ε, καταπολέμησης τρομοκρατίας. Έχω ε, θύματα από την οικογένειά μου εσείς δεν έχετε υποστεί διώξεις ποτέ. Δεύτερον, μόλις επέστρεψα από την Μόρια αγαπητέ και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτά που είδα εκεί στο στρατόπεδο, στο κέντρο υποδοχής ε, εκεί είναι απολύτως απαράδεκτα υπό την ε, οπτική των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων για τις αξίες που θέλουμε να έχουμε εμείς ως Ευρωπαίοι σε όλα αυτά που κάνουμε, διότι το κέντρο εκεί το να περάσει κανείς ένα χειμώνα ή ένα φθινόπορο με τις απάνθρωπες συνθήκες, χωρίς πόσιμο νερό, τρεχούμενο, με διακοπές υδροδότησης, με παιδιά που βρίσκονται εκεί μήνες και μήνες, με τα τραύματα που αφήνει στους ανθρώπους αυτούς και στα παιδιά η, διαβίωσή τους εκεί, η παραμονή τους εκεί, αυτό είναι κάτι που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ δεν είμαι καθόλου ακραία. Δεν είμαι εξτρεμίστρια. Προσπαθώ να δω τα πράγματα λογικά. Αλλά εδώ μιλούμε για ιδεολογικό εξτρεμισμό. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε λογικά και με συνέπεια να εφαρμόζουμε την ομοθεσία και το να διατηρούμε ανθρώπους σε κέντρα τέτοια περνώντας μήνες και μήνες για να, δούμε, για να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε μαζί τους, για να δούμε πώς θα διαβιβάσουμε τα στοιχεία τους και τους φακέλους τους και, και στο μεταξύ να μένουν όλο αυτό το διάστημα σε τέτοια κέντρα παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Και εγώ την αναφορά αυτή την απέστειλα στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για να δουν αν αυτά είναι τα πρότυπα που πρέπει να αποδεχόμαστε εμείς ως πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα επιχειρήματα. Αν, η αν τα πράγματα στη Λιβύη έχουν, όπως λένε, τότε δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια για κάτι που προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Επιστρέφω λοιπόν επιχειρήματα σε αυτά που λέτε. Μη λέτε αβάσιμα πράγματα. Ε, ο πρόεδρος. Κοιτάξτε, εγώ το μόνο που σας ζητώ ε, είναι να μην, ε, να μην πέφτετε στην παγίδα της πρόκλησης, συνάδελφοι. Δεν χρειάζεται να απαντούμε σε όλες τις προκλήσεις. Ο καθένας έχει τις απόψεις του, όχι απολύτως σεβαστές, αλλά εμπασιτός τις απόψεις του. Ο κύριος Κώστερ. Εγώ, λέει ο κ. Κέστερ, επιθυμώ να τονίσω πρώτα ότι αισθάνομαι απόλυτη αλληλεγγύη με τις ε, διασωστικές οργανώσεις. Η υποστήριξη όσο, όσο γίνεται περισσότερων ευρωβουλευτών, όσο είναι δυνατόν δηλαδή, είναι αναγκαία. Και προέρχεται και από μια έκφραση επιθυμίας των ανθρώπων που φτιάχνουν αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση και που οι χώρες αυτή τη στιγμή αποτυγχάνουν να υλοποιήσουν μια πολιτική που να υπερασπιστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό θεωρώ ότι οι διασωστικές οργανώσεις δρούν μεταξύ άλλων και υπέρ της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι η ιδέα ότι η εφαρμογή αυτών των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των ανθρώπινων αξιών, ότι αυτά τα πράγματα δεν εφαρμόζουμε απέναντι στους πρόσφυγες, σημαίνει μεταξύ άλλων ότι τις αξίε αυτέ τι αμφισβητούμε και εμεί οι ίδιοι για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι τι αμφισβητούμε όχι μόνο στη στάση μα απέναντι στους πρόσφυγε, αλλά και μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν οι ανθρώπινες αξίε έρχονται σε τέτοια σύγκρουση με την πραγματικότητα, όπω γίνεται τώρα, τότε εν τέλει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση αμφισβητείται. Αυτό πρέπει ε, να το έχουμε απόλυτα καθαρά στο μυαλό μα. Και παρόλα αυτά να πω κάτι για αυτό που λέχθηκε προηγουμένως. Τα ανθρώπινα δικαιώματα ισχύουν υπέρ όλων, όχι μόνο υπέρ των Ευρωπαίων. Είναι, πώς να πω, το βασικό επίτευγμα της σύγχρονης εποχής. Και να πιστεύουμε ότι μπορούμε να αφήσουμε παιδιά, ανήλικους, γυναίκες, γέρους να πνίγονται στην Μεσόγειο μόνο και μόνο διότι έρχονται, λέει, να εκμεταλλευτούν τα συστήματα κοινωνική ασφάλειας, εγώ το θεωρώ αυτό πραγματικά απολύτω απαράδεκτο. Και αυτού του είδου η νοοτροπία και αυτού του είδους η συμπεριφορά θα καταστρέψει εν τέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται να περάσει. Σύπερ, το Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σμιτ και τον κύριο Μεχρατόμ που είναι σήμερα εδώ, αλλά και να τους ζητήσω συγγνώμη για αυτά που άκουσαν. Θα συμφωνήσω με τη συνάδελφό μου Κρίστα ότι η ποινικοποίηση της διάσωσης, η εκ των προτέρων καθολική καταδίκη όλων των προσώπων που προσέρχονται μεταναστών ή προσφύγων δεν αποτελεί μονάχα παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και παραγνωρίζει τη δυστυχία πολλών ανθρώπων, αλλά θέτει σε κίνδυνο και την ίδια την Ευρωπαϊκή Συνοχή και αντιβαίνει καθαρά το κράτος δικαίου, της ανθρώπινης αξίες και ρίχνει νερό στον μήλο των εξτρεμιστών. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, ο πολιτισμός όλων των χωρών μελών, εδώ και αιώνες είναι ανάμεικτος, σύμμικτος ε, πολιτισμός μέσα από όλου τους αιώνε όλοι οι Ευρωπαίοι μετακινήθηκαν, καμιά φορά με το ζόρι, καμιά φορά με τη θέλησή του και έτσι έχουν μεταφέρει τον πολιτισμό τους από μια χώρα στην άλλη. Και σήμερα βρίσκουμε σε πολλές χώρες της Ευρώπης τα απομεινάρια του τουρκικού και του αραβικού πολιτισμού. Είμαστε μια ανάμεικτη ήπειρο και όλοι φέρουμε τη σχετική ευθύνη. Η ποινικοποίηση καταστρέφει όχι μόνο τις δικές μας αξίες, αλλά συμπεριφερόμαστε περιφρονητικά και απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να ζητήσουν τη βοήθειά μας. Δράμα για αυτούς που έρχονται, αλλά και δράμα για αυτούς που ήδη είναι εδώ παροιμήν. Αν αύριο πάψουν να έρχονται οι μετανάστες, σε ποιους θα στραφεί το μίσος που υπάρχει και βράζει. Ότως ή άλλως, η αλλω η απορριψη των μεταναστών είναι κακό από μόνη της, αλλά αύριο θα στραφεί και κατά πολλών άλλων και θεωρώ ότι όλοι καλά θα κάνουμε ε, για το ερώτημα πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή, να επανέλθουμε στις θεμελιώδεις αξίες, διάσωση των ανθρώπινων ζώων, να δεχτούμε τους ανθρώπους με συνθήκες αξιοπρέπειας. Και ναι, βέβαια, δεν μπορούμε να υποδεχθούμε 60 εκατομμύρια πρόσφυγες από όλο τον κόσμο εδώ, παροιμήν, αλλά ούτε θα έρθουν και τόσα πολλά, ούτε είναι δυνατόν. Αν θέλουμε όμως μακροπρόθεσμα να μειωθεί ο αριθμός των προσφύγων, όχι μόνο αυτών που έρχονται προς εμάς, αλλά και όλων συνολικά. Οι αριθμοί των προσφύγων, αυτών δηλαδή των προσώπων που νιώθουν αναγκασμένα να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους για κάποιο λόγο. Τότε πρέπει να αλλάξουμε όχι μόνο το σύστημα ασύλου, πρέπει να αναζητήσουμε νόμιμες οδούς μετανάστευσης, αλλά πρέπει και να σταματήσουμε να ποινικοποιούμε τις προσπάθειες των διασωστών και χρειαζόμαστε και άλλου είδους συνεργασία με χώρες προελεύσεως και με τρίτες χώρες. Και εκεί πρέπει να στρέψουμε τις προσπάθειές μας και όχι σε μια δίθεν ερμητική φραγή απέναντι σε άλλες χώρες και υπήρους του κόσμου. Η Ευρώπη δεν καταδυναστεύει τον κόσμο, αλλά συνεργάζεται με άλλους για να βρει κοινέ λύσεις. Ευχαριστώ, κύριε Σπινέλη. Ευχαριστώ, Αντώνιο. Η συζήτηση που έγινε μεταξύ δύο βουλευτών για το θέμα της μετανάστευσης και της ε, τρομοκρατίας δεν είναι συζήτηση μεταξύ απόψεων που απέχουν την πραγματικότητα. Αυτό που αναφέρθηκε για τη σχέση μεταξύ μετανάστευσης και τρομοκρατίας είναι αυτό που λένε οι κυβερνήσεις ε, μεταξύ τους και η Ιταλική κυβέρνηση πρώτη και καλύτερη. Σας αναφέρω μόνο τι έλεγε ο αντινάβαρχος Δεφελίτσε που, ασχολ, που μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν ε, υπεύθυνο για την ε, Σικελία, ο οποίος συστήνει μια ασφαλή λύση για το πρόβλημα των μεταναστών που συνίσταται στο εμπάργο, στον αποκλεισμό των παράκτιων ε, περιοχών, ε, των παράκτιων ζωνών της Λιβύης, ε, επικαλούμενο στο άρθρο 33 <clears throat> του κώδικα διεθνούς ναυσιπλοείας για την, για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η ιδέα λοιπόν αυτή δεν είναι ιδέα μόνο ενός βουλευτή αλλά και των κρατών μελών της Ένωσης. Μια άλλη κυρίαρχη ιδέα σε πολλά κράτη της Ένωσης και στην Επιτροπή είναι ότι η διάσω, το Search and Rescue, η διάσωση στη θάλασσα, όχι το Search and Rescue από τις ΜΚΟ, αλλά γενικά η διάσωση στη θάλασσα είναι λάθος, διότι είναι επικίνδυνο να διασώζεις άτομα στη θάλασσα. Η, ζωή των ανθρώπων θεωρείται κάτι επικίνδυνο που πρέπει να αποφεύγεται, έστω και αν αυτό οδηγεί στην, στον πνιγμό τους. Αυτό το λέμε το, τώρα στο τέλος της θητείας όπου τα λέμε πέρα πράγματα λέμε εδώ και τέσσερα χρόνια. Κάτι άλλο που βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα και που γνωρίζουν πολύ καλά οι μη κυβερνητικέ οργανώσει κατά την άποψή μου είναι ότι τα προβλήματα που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν στη θάλασσα, στη θάλασσα εφαρμόζεται ο νόμος, διασώζονται αυτοί που πρέπει να διασώζονται και περιμένουν να γίνεται πολιτική στη θάλασσα. Δηλαδή την πολιτική που πρέπει να γίνεται στην ε, στεριά την κάνουμε στη θάλασσα, χρησιμοποιώντας τους μετανάστευς ως όμοιρους για 30-60 μέρες για να πετύχουμε κάτι στην Ευρώπη, μια μετεγκατάσταση. Αυτό είναι ένα από τα πιο επέσχυντα και σκανδαλώδη πράγματα που συμβαίνουμε. Η ανάμειξη του διεθνούς δικαίου και των, πολιτικών, των κρυφών πολιτικών δράσεων, η, η διεθνής νομοθεσία, το διεθνές δίκαιο εξαφανίζεται παντελώς. τελειώνω πάντα στην, στο σκεπτικό ασφάλεια, τρομοκρατία. Έχουμε πολλά, πολύ λίγα παιδιά στην Ευρώπη, αυτό είναι πρόβλημα, αλλά ταυτόχρονα αφήνουμε τον κόσμο να πεθαίνει στη θάλασσα. Τώρα, το άλλο ζήτημα είναι το καλοκαίρι. Έχουμε εκλογές, ευρωεκλογές και ταυτόχρονα καλοκαίρι. Αναγγελία μεγάλων εισβολών, μεταναστευτικών εισβολών ε, στην Ευρώπη από ό,τι παράλογα και ψεύτικα ε, παράλογες και ψεύτικες ειδήσει μπορείτε να φανταστείτε. Βέβαια δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Θυμίζω ότι το 90% των μεταναστών ανά τον κόσμο βρίσκονται στην Αφρική, την Ασία και τη Νότια Αμερική. Στην Ευρώπη είναι το 2%. Σκεφτείτε το λίγο πιο ξεκάθαρα. Ευχαριστώ. Sentiamo ε, ας ακούσουμε τώρα την ε, Rettet, που είναι μια μη Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για να τοποθετήσω λίγο αυτά που είπε ο κύριος προηγουμένως. μπορέσαμε, γιατί λέει ότι διασώζονται διάφοροι κτλ. Ξεκίνησε από ένα Ολλανδικό think tank το οποίο μάλιστα παρακολουθείται από τις μυστικές υπηρεσίες, διότι έχει βαθιά εθνικιστικό χαρακτήρα. Όποιο λοιπόν απευθύνει τέτοιες κατηγορίες, εδώ ή έξω ή και στο living room του, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να συνεργάζεται με ε, εθνικιστές του χειρίστου είδους. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι οποιαδήποτε μη κρατική οργάνωση έκανε κάτι λάθος, διότι απολύτως τίποτε λάθος δεν έκαναν. Τόσο απλά είναι μερικές φορές τα πράγματα. Avete qualcosa da rispondere? Έχουμε κάτι να απαντήσουμε, λέει ο Πρόεδρος, στις παρατηρήσεις αυτές. No, basta. I've, I've nothing to add to... Ε, πρόεδρε, δεν έχω να προσθέσω εγώ κάτι. Okay. I have a right to answer for, for, for... Έχω το δικαίωμα να απαντήσω, Πρόεδρε. Ε, δεν είναι διάλογος αυτός ε, μεταξύ σας, λέει ο πρόεδρος. Ε, Οπότε τι είναι, λέει ο μιλητής. Γιατί έτσι αποφάσισα εγώ. Έτσι αποφάσισα εγώ, λέει ο πρόεδρος. Δεν είναι συζήτηση, δεν είναι διάλογος. Και τι είναι. Τι είναι, πρόεδρε. Σταματήστε, λέει ο πρόεδρος. Θα περάσουμε τώρα στο δεύτερο σημείο για τις διασώσεις, επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα και το διεθνέ δικαίο. Όταν μιλούμε για τη δραστηριότητα των ΜΚΑΟΜΚΡΟΝ στην Μεσόγειο, πέραν του ανθρωπισμού, οι επιχειρήσεις διάσωσης ε, στη θάλασσα πρέπει να υπακούει και στις ε, διεθνείς της διατάξεις, μάλλον του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Έχουμε εδώ τον κύριο Νταβίδ από το Πανεπιστήμιο ε, των Βρυξελών, που θα μας βοηθήσει, θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου σχετικά με τις διατάξεις αυτές και σας δίνω μέσα το λόγο, κύριε Νταβί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι μπορώ να μιλήσω στα γαλλικά, λέει ο μιλητής. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι θαυμάσιο. Είναι θαυμάσιο, λέει ο μιλητή στα αγγλικά. Πού μπορώ να μιλήσω στα γαλλικά. Και συνεχίζει ο μιλητής στα γαλλικά. Είναι ανακούφιση που μπορώ να μιλήσω στα γαλλικά καθότι είμαι και ακτιβιστής κατά του γλωσσικού υπερελεγισμού των Αγγλικών. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε στην ε, συνάντηση αυτή. Αυτά που θέλω να πω είναι αρκετά απλά και νομίζω ότι οποιοδήποτε φοιτητή στο τρίτο έτος του, της νομικής, στο δίκαιο, θα μπορούσε να σας εξηγήσει. Έχω μία παρουσίαση σε τέσσερα τμήματα. Πρόεδρε, εάν μακρηγορήσω, μην διστάσετε να με διακόψετε. Ήθελα να αναφερθώ καταρχάν για την υποχρέωση παροχής βοήθειας. Δεύτερον, για τις ποινικέ διώξεις της παροχής αυτής βοήθειας. Τρίτον, για τις ε, δικαστικές προσφυγές που γίνεται να υπάρχουν και τέταρτον για την υποχρέωση της δικαιούς κατανομής του άχθους υποδοχής των προσφύγων. Καταρχάς λοιπόν για την ε, συνδρομή, την παροχή βοήθειας. Αυτή η συνδρομή, η υποχρέωση μάλλον της συνδρομής ανθρώπων που κινδυνεύουν αναφέρεται στο άρθρο 98 στο άρθρο 98, το λέω βελγικά αλλά δεν πειράζει, 98 λοιπόν, τη σύμβαση που λέγει ότι όλες οι χώρες με σκάφος, με πλοίαρχο και σκάφος που λειτουργεί υπό τη σημαία του θα πρέπει να διασώζουν ανθρώπους που κινδυνεύουν στη θάλασσα. Αυτό είναι αρκετά σαφές πιστεύω. Δηλαδή, το να βοηθούμε ανθρώπους που κινδυνεύουν στη θάλασσα ή σκάφη τα οποία κινδυνεύουν να βυθιστούν είναι από, τα, από τις βασικότερες διατάξεις της σύμβασης Μοντεγκόμπε και το να μην το πράξει κανείς αυτό, το να μην παράσχει συνδρομή <clears throat> θα σήμαινε ότι η χώρα της οποίας το σκάφος μιας που δεν θα το έκανε θα διέπρατε ένα αδίκημα υπό το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ένα δεύτερο στοιχείο, πάντα σε αυτό το πλαίσιο υποχρέωσης συνδρομής, μετά τις τελευταίες παρατηρήσεις που ακούσαμε τις παρεμβάσεις, τίθεται το ερώτημα μπορούμε να σταματήσουμε στα ανοιχτά της θάλασσας ένα σκάφος το οποίο μεταφέρει πρόσφυγες. Όχι. Και εδώ δεν αναφέρομαι στη Διεθνή Σύμβαση του Δικαίου τη θάλασσα, Αναφέρομαι στην συνθήκη της Γενέβης του 1951 για το καθεστώς προσφύγων. Την οποία ε, τροποποιεί το πρωτόκολλο του 67 και που λέγει <clears throat> ότι όλοι αυτοί που διαφεύγουν από τη χώρα τους γιατί υφίστανται διώξεις ε, εθνικές, θρησκευτικέ, πολιτικές ή άλλες μπορούν να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες. Και επομένω αποτρέποντας από τους ανθρώπους αυτούς να ασκήσουν το δικαίωμά τους δηλαδή να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες είναι επίσης αδίκημα διότι δεν αναγνωρίζουμε ένα δικαίωμα που αναφέρει στο πρώτο άρθρο της η συνδίκη της Γενέβης του 1951. Αυτά για την υποχρέωση συνδρομής. Δεύτερον τώρα. Οι διώξεις. Η ποινική δίωξη που μπορεί να ασκηθεί προς τις οργανώσεις, τις ενώσεις, της μη καπαόμικρων που παρέχουν συνδρομή σε Η άσκηση δίωξης, η κατηγορία προς τους εκπροσώπους των ενώσεων αυτών, η ποινική δίωξη, θα έπρεπε να βασίζεται στις διατάξεις που μόλις ανέφερα και όπως γνωρίζετε το διεθνές δίκαιο παραπέμπει στην νομοθεσία των χωρών που ενέχονται και επομένως ένας δικαστής θα έπρεπε εδώ πρώτα απ' όλα να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο. Και λέγω το να μην συνδράμουμε ανθρώπους που, που, μόλις, ε, ε, που βρίσκονται στη θάλασσα μετά από ναυάγιο θα ήταν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και μία μη καπαόμικρον που θα εδιώκετο επί τη βάση αυτή θα μπορούσε να στραφεί σε οποιονδήποτε καλό δικηγόρο ώστε να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο και η υποχρέωσή της να συνδραμεί. Εάν μάλιστα <clears throat> ελάμβανε χώρα μια τέτοια δίεξη, τότε θα υποχρεούται το κράτος να αναγνωρίσει τις διατάξει του εθνούς δικαίου και σχετικά με τις προσφυγές δικαιοσύνη, οποιαδήποτε ποινική δίωξη θα μπορούσε να ασκηθεί κατά ανθρώπων οι οποίοι ασκούν αυτήν την υποχρέωση συνδρομή στην ανοιχτή θάλασσα, θα μπορούσαν να παραπέμψουν στο άρθρο 98 της Σύμβασης Μοντεγκομπέ που μόλις ανέφερα πριν. Επίσης θα μπορούσαν να αναφερθούν στο πρώτο άρθρο τη ε, συνθήκη για τους Πρόσφυγες της Γενέβη του 1951. Και θα μπορούσε να φανταστεί κανείς αρκετά εύκολα ότι η χώρα από την οποία προέρχονται οι άνθρωποι αυτοί που κινδυνεύουν και δεν τους παρέχεται συνδρομή ή που αποτρέπουμε από κάποιους να τους παράσχουν συνδρομή, η χώρα αυτή θα μπορούσε να ε, προστατεύσει διπλωματικά τους ανθρώπους αυτούς και να αναλάβει δράση κατά του κράτους εκείνου που θα ήταν αντίθετο προς τη διάσωση αυτή στη θάλασσα ή προς την ελεύθερη διέλευση των ανθρώπων αυτών που θέλουν απλώς να αναγνωριστεί το δικαίωμά τους να είναι πρόσφυγες. Δηλαδή έχουμε διατάξεις σχετικά με την δικαστική αρμοδιότητα, δυνατότητα προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο, στα Ηνωμένα Έθνη ή και μέσω ερωτήματος που θα μπορούσε να απευθύνεται στο δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και το οποίο θα μπορούσε και αυτό να έχει αρμοδιότητα επί των θεμάτων αυτών και να παραπέμπει σε αντίστοιχε διατάξει των διεθνών συνθήκων. Το τέταρτο σημείο που ήθελα να θίξω, να εξηγήσω, ήταν η υποχρέωση αλληλεγγύης, για να το πούμε έτσι. Και επίσης η δίκαιη κατανομή του άχθους της ε, υποδοχής ε, των, προσφύγων. Έχουμε το άρθρο 80 της Ειδίκης Λισαβόνας για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προβλέπει ότι όλες οι χώρες οφείλουν ισότιμα να παρέχουν βοήθεια η μία στην άλλη και να κατανέμουν σωστά και δίκαια το άχθος της υποδοχής των ανθρώπων αυτών. Μπορούμε να φανταστούμε επίσης λοιπόν εξίσου εύκολα ότι ένα κράτος θα μπορούσε να αναλάβει δράση να προσφύγει κατά άλλου κράτους στο δικαστήριο στο Λουξεμβούργο κατά άλλου κράτους που δεν σέβεται, που δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 80 της Συνθήκης για Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει γίνει ακόμα κάτι τέτοιο, αλλά με εκπλήσει θα μπορούσε ωραιότατα να γίνει κάτι τέτοιο, μια τέτοια προσφυγή δηλαδή. Και δεν μιλούμε μόνο για μια υποχρέωση η οποία αναφέρεται στο άρθρο 80 της συνθήκης Λισαβόνας. Βρίσκουμε το ίδιο, την ίδια διάταξη, στην παράφορα 133 του τελικού εγγράφου του 2005 που ενέκρινε η Ολομέλεια των Ηνωμένων Εθνών στο ψήφισμα 60 1 που λέει ακριβώς το ίδιο. Αναφέρει αυτήν την υποχρέωση δίκαιης ισότιμης κατανομής του άχθους, δηλαδή αλληλεγγύη μεταξύ όλων των χωρών, σχετικά με την υποδοχή των προσφύγων. Επομένως, δεν είναι ιδιαίτερα περίπλοκες οι διατάξει του δικαίου, αρκεί να το εφαρμόζει κανείς. Έχουμε τα διεθνή δικαστήρια, έχουμε πολλά μέσα εργαλεία στη διάθεσή μα, αλλά δυστυχώς συχνά οι νομικοί δεν χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά που έχουν στη διάθεσή τους. Αρκεί κανεί να ανοίξει τα βιβλία, να δει τι διατάξεις, αυτές δηλαδή που εντάχει σας επεσήμενα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Κλοντ. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. δεν ήταν σαν και εσάς οι καθηγητές νομικής που είχα όταν σπούδαζα νομική. Μ' άρεσε αυτό που είπατε ότι τα νομικά εργαλεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Δεν το έκαναν αυτό. Τελειώνουμε την εκδήλωση αυτή για το βραβείο Ζαχάροφ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τρει από του διοργανωτέ, τρει από τι μη κυβερνητικέ οργανώσει που είναι πλέον δραστηριε στη Μεσόγειο, Open Arms, ε, ε γιατροί χωρίς σύνορα και ΝΟΑΣ. Ο Ρικάρντο Γκάτι από το Open Arms έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω Ιταλικά. για να μιλήσουμε για τις μελλοντικέ προκλήσεις στην κεντρική Μεσόγειο, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς να δούμε με κριτική προσέγγιση αυτό που συμβαίνει στην κεντρική Μεσόγειο τώρα. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Όπως αναφέρθηκε και εξηγήθηκε από τους διάφορους ομιλητές ε, σήμερα, η κατάσταση στο πλαίσιο της οποίας ε, βιώνουμε τη διαδικασία αυτή οι μη κυβερνητικέ οργανώσει εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια είναι ακόλουθη. Καμία μη κυβερνητική οργάνωση διάσωση στη θάλασσα δεν έχει ε, μια σειρά δράσεων καταστολή εις βάρος τους εκτός της, ε, εκτός της ε, νομοθεσίας με, πολιτικές, με πολιτικούς στόχους καταχρήσεων, δράσεων ε, δυσφήμισης, ε, ψευδής, ψευδούς ενημέρωσης και συστηματικής καταγγελίας των ίδιων των ΜΚΟ. Είναι ανησυχητικό να βλέπουμε πως ε, προχωρούν κατηγορίες ατιμόρυτα για επιθέσεις, ένοπλες επιθέσεις εις βάρος των σκαφών των ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ιταλία και τη Γαλλία που, από την Ευρώπη που πυροβόλησε και συνέλαβε εμένα τον ίδιο σε κάποιες περιπτώσεις. Την υποστήριξη που δίνουν ε, τα κράτη της Ένωσης στην ακτοφυλακή της Λιβύης. Ε, η επίθεση εις βάρος ε, των σκαφών μας από σκάφη χωρίς νομική υποστήριξη που παρεμπόδισε πρόσβασης στα λιμάνια της Ιταλίας χωρίς μια σειρά περίπλοκων ε, απαιτήσεων χωρίς ε, και ανιδιολόγητων απαιτήσεων που οδηγούν στην ε, μη εφαρμογή των κανόνων που θα έπρεπε να σέβονται τα θεσμικά όργανα της Ιταλίας. Η, τροφο, η έλλειψη, η δυσκολία τροφοδοσίας των σκαφών μας οδηγώντας τα σκάφη σε καταστάσεις αδυναμίας αποβίβασης των ατόμων σε ασφαλή λιμένα. Έρευνες και πολλαπλές από πλευράς των Ιταλικών αρχών που ωστόσο εδώ και χρόνια δεν οδήγησε σε καμία καταδίκη. Άρνηση χορήγησης άδεια προσόρμησης ή ε, κατακράτησης καυσίμων, σκαφών ή αεροσκαφών. Έλλειψη ενημέρωσης για το τι συμβαίνει τόσο στην Κεντρική Μεσόγειο και στη Λιβύη. Μέχρι σήμερα είναι αδύνατο να ξέρουμε πόσα άτομα έχουν πεθάνει, πόσα άτομα έχουν ε, συλληφθεί και επιστραφεί στα κέντρα, στα κέντρα κράτησης, που, στα, στα, στα στρατόπεδα συγκέντρωση που συνεχίζουν να καλούμε κέντρα κράτησης. Δράσεις αυτές ε, ε, επινοήθηκαν και οργανώθηκαν με σαφή στόχο να καταστήσουν αυτό που συμβαίνει στην Κεντρική Μεσόγειο και κατά συνέπεια αυτό που συμβαίνει στη Λιβύη αδύνατο να γίνει κατανοητό και να γίνει γνωστό, ούτω ώστε να δημιουργηθεί ένα ρεύμα σκέψης που θα μπορούσε να αντισταθεί στις πολιτικές εξωτικερίκευσης των ε, εξωτερικών μας συνόρων, που, με πολιτικές που δεν θέτουν στο κέντρο τον άνθρωπο και που οδηγούν σε σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Είναι προφανές ότι όλα αυτά επιβάλλουν ε, σοβαρές ε, σκέψεις στα δικά μας θεσμικά όργανα, τα οποία όλα αυτά τα χρόνια έχουν στόχο να απομακρύνουν τη μαρτυρίες ε, των μαρτύρων και που οδηγούν στην, στην συνεχή παρουσίαση των ψευδών ειδήσεων η βάρος των μεταναστών. Μέχρι σήμερα οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις που βρίσκονται στην κεντρική Μεσόγειο βρίσκονται είτε στην ανάγκη να εγκαταλείψουν την υποστήριξη, την τα, τις προσπάθειές τους ή να επιστρέψουν στα λιμάνια χωρίς καμία υποστήριξη από τα κράτη και με κίνδυνο τη ζωή τους. Ε, βεβαίως η κατάσταση ποικίλει από χώρα σε χώρα, από που προέρχονται και από την ε, υποστήριξή τους. Ωστόσο, η υποστήριξη των, ε, των προσπαθειών διάσωσης από πλευράς μας έχονται σε αντίθεση και με τις πολιτικές που, που δίδονται εις βάρος των, ε, της ακτοφυλακής της Οι προσπάθειες των αρχών να μεγιστοποιήσουν τους σπόρους ούτως ώστε να καταστήσουν δύσκολη την ε, αποβίβαση των ε, ε, προσφύγων σε ασφαλή λιμένα επιδεινώνεται ενώ τα κράτη κρύβονται πίσω από το ότι οι αρμόδιες αρχές συντονισμού της διάσωσης στην περιοχή αυτή γίνονται ε, εκτός ευρωπαϊκών συνόρων. Στην πραγματικότητα όλα αυτά γίνονται από παρότι ε, στη, η ακτοφυλακή της Λιβύης ουδέποτε απαντά στα τηλέφωνα. σήμερα το πρωί, οκτώ από τα 8 τηλέφωνα που είχαμε για την ακτοφυλακή απάντησε το ένα και ο άνθρωπος που απάντησε δεν ήξερε αγγλικά. Μπορείτε να φανταστείτε ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει χωρίς την υποστήριξη των ΜΚΟ σε καθημερινή βάση που έχουν στόχο να προστατεύσουν τη ζωή των ανθρώπων και τα δικαιώματά τους στην θάλασσα. Μετά την διάσωση το δεν επιτρέπεται η αποβίβαση στα Ιταλικά λιμάνια. Αυτό το λένε, Ιταλικές, το λένε Ευρωπαϊκές Αρχές που επιμένουν ότι πρέπει τα άτομα αυτά να επιστραφούν στη λιμή δείχνοντας είτε άγνοια του διεθνούς δικαίου είτε αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή. Μετά την, προς την διάσωση των ατόμων, τα σκάφη μας παραμένουν εκτός ε, χωρικών υδάτων για, για πολλές μέρες ε, υπό την πίεση των Ιταλικών αρχών και οι φυστάμενες περίεργες διαδικασίες όπως η Ισπανική κυβέρνηση που ε, τονίζει ότι η παραμονή στη θάλασσα σε ανοιχτό στο, στα διεθνή ύδατα για πολλές μέρες ενός σκάφου οδηγεί σε παραβίαση των δικαιωμάτων των ανθρώπων. Θέλω να υπενθυμίσω ότι το δικό μας σκάφος, το Open Arms, είναι τυπικά σκάφος ε, παρατήρησης και διάσωσης όπως ακριβώς τα σκάφη που, έχουν, που έχει η Ιταλική, η Ισπανική ε, ακτοφυλακή. Η είσοδος στο λιμάνι, στα λιμάνια καθυστερεί για μέρες μετά από έρευνα των εισαγγελιών και ε, με, επι, με επιβάρυνση των Κλείνω. Η προσπάθεια των μη κυβερνητικών οργανώσεων εφαρμόσουν την αλληλεγγύη στη θάλασσα ε, αυτή τη στιγμή ε, αναστρέφεται παντελώς. Οι πολιτικοί δεν γνωρίζουν ή δεν θέλουν να γνωρίζουν τι σημαίνει κακομεταχείριση των ανθρώπων και αντιμετωπίζουν τους ε, μετανάστες και πρόσφυγες με τρόπο που αποδείχνει, που αποδεικνύει ότι δεν σέβονται καθόλου την ανθρώπινη ζωή. Η ερώτηση που θέτω, ποια κοινωνική λογική κατευθύνει τις, τους θεσμούς που μπορούν να επιτρέπουν στις κυβερνήσεις να εφαρμόζουν ατιμωρητή σειρά πράξεων εις βάρος των δικαιωμάτων των ανθρώπων, εις βάρος της ζωής των ανθρώπων και εις βάρος των ε, χωρών μας όταν βλέπουμε ότι οι δράσεις ε, φανατικών αυξάνονται. Αυτό που θέλω να πω στο τέλος είναι ότι έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι όλα αυτά, όλες αυτές οι κατηγορίες είναι ψευδείς. Ψευδείς είναι και, όλες οι και όλα τα άλλα fake news εις βάρος των μη κυβερνητικών οργανώσεων που κάνουν διάσωση στη θάλασσα, που μέσω των ε, μέσω των, ε, των ε, ραδιοφωνικών μηνυμάτων είχαν οδηγήσει σε αποκλεισμό ορισμένων σκαφών. Πώς μπορεί να επιβιώσει μια τέτοια κοινωνία. Τι κάνουμε, πώς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το μέλλον μας. Ευχαριστώ. Thank you very much, uh, Ricardo. <clears throat> Uh, Σας ευχαριστώ πολύ, Ρικάρντο. Πριν λίγους μήνες, μήνες πέρασα από τη Λιβύη λίγες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Κάποιες, μια από αυτές ήταν ε, των γιατρών χωρίς σύνορα και πολύ ευχαρίστως ε, θα δώσουμε το λόγο στην κυρία για να μιλήσει ακριβώς για τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Είμαστε ακόμα παρόντες σε Τρίπολη, Μισουράτα και Χόμς που εκεί γίνονται μερικές αποβιβάσεις τώρα, οι πιο πρόσφατες δηλαδή, και έχουμε κάποιες μαρτυρίες. Θα προσπαθήσω να μην μιλήσω μόνο για μαρτυρίες και συναισθηματικά φορτισμένες ιστορίες, αλλά θα σας δώσω και συγκεκριμένα νούμερα. Και στην παρουσίασή μου μπορώ να την περιορίσω σε ένα λεπτό. Δεν υπάρχει επαρκής βοήθεια, προστασία και ούτε εναλλακτικέ επιλογές στην ένταση και ούτε και υπάρχει και καμιά άλλη δυνατότητα από το να επιστραφούν στις πατρίδες τους. Όποιος έχει περάσει από αυτά τα κέντρα κράτησης γνωρίζει ότι αν δεν θέλει κάποιος να γυρίσει πίσω εθελοντικά, θα πρέπει να έχει πάρα πολλού σοβαρούς, λόγους για να μην πάει. Με το παράδοξο ότι πιο, τα πιο ευάλωτα άτομα σήμερα είναι αυτά τα οποία έχουν παγιδευτεί στην ΒΗΗ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, βοήθεια σε τόπους αποβίβασης, θεωρητικά τα Ηνωμένα Έθνη και οι εταίροι τους είναι σε 12 σημεία αποβίβασης. Οι γιατροί χωρίς σύνορα όχι στην Τρίπολη, είμαστε όμως τώρα στη Μιζουράτα και στην Χόμς και προσπαθούμε να καλύψουμε και άλλα σημεία, αλλά δεν έχουμε συστηματική παρουσία. Μόνο όταν μας δέχονται να πάμε ή όταν μας ζητήσουν να πάμε. Δεν μπορούμε αυτομάτως να πάμε, δηλαδή όταν γίνεται μια αποβίβαση. Ακόμα και με την παρουσία μας ωστόσο εκεί και ε, μαζί με το διεθνές προσωπικό, η ικανότητά μας να βοηθήσουμε είναι πολύ περιορισμένη. Μπορούμε δηλαδή να προσφέρουμε κάποιες ε, πολύ βασικές πρώτες βοήθειες και δεν έχουμε λόγο καθόλου για το πού θα μεταφερθούν τα πρόσωπα αυτά. Το πολύ που μπορούμε να κάνουμε είναι για τις ιατρικές παραπομπές, για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε πραγματικά άσχημη κατάσταση. Στις πιο πρόσφατες αποβιβάσεις που έχουμε καταστεί μάρτυρες είδαμε πολύ ψηλό αριθμό ανθρώπων ε, που πάσχουν από ασυτεία. Και αύριο θα μιλήσω για την ασυτεία σε ένα από τα κέντρα κράτησης. Όμως αυτό δεν συμβαίνει λόγω της παραμονής τους στη θάλασσα, αλλά διότι πέρασαν μακρές περιόδους με πολύ κακή σύντηση σε κέντρα επίσημα ημί. Με πάρα πολύ περιορισμένη πρόσβαση σε διατροφή. Έχουμε και σοβαρές ε, ιατρικές επιπλοκές. Πέντε άτομα χρειάστηκε να παραπέμψουμε μεταξύ αυτών και ανηλίκους, ένα παιδί 15 χρονών από τη Σομαλία που μάλιστα απεβίωσε. Και επίσης πολλές γυναίκες και παιδιά και έγκυες γυναίκες. Και είχαμε και την περίπτωση μιας γυναίκας πολύ προχωρημένη εγκυμοσύνης, την έστειλαν στο κέντρο ε, κράτησης γέννησε, μπορέσαμε να την παραπέμψουμε σε νοσοκομείο, σε ιατρικό κέντρο δηλαδή, και μετά από τον τοκετό χρειάστηκε να επιστρέψει στο κέντρο κράτηση. Δεν μπορούμε δηλαδή να του διακινούμε όλου. Και δεν μπορέσαμε να επιτύχουμε στη γυναίκα αυτή να μην επιστραφεί. Μπορέσαμε τελικά μάλλον, ήταν πάρα πολύ δύσκολη και δυσκίνητη η διαδικασία αυτή. Και τα καταφέραμε και με άλλε τέσσερι γυναίκε. Αυτό το μετράμε ω τεράστια επιτυχία. Να μπορέσουμε δηλαδή τέσσερι γυναίκε με μωρά. Να τα βγάλουμε, να τις βγάλουμε από τα κέντρα κράτησης είναι τεράστια επιτυχία και η οργάνωσή μου είναι πάρα πολύ ε, ευχαριστημένη που το πέτυχε. Σε ό,τι αφορά την παροχή προστασίας. Όπως είπα, βοήθεια μπορούν να προσφέρουν πολύ περιορισμένη. Για προστασία, όταν αποβιβάζονται οι άνθρωποι, επισήμως πρέπει να πάνε σε κέντρο κράτηση, επίσημο κέντρο κράτησης. Όμως οι διακινητές είναι επίσης παρόντες Στι αποβιβάσεις, ακόμα και όταν είμαστε και εμεί παρόντες εκεί. Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνονται όλοι όσοι αποβιβάζονται. Έχω κάποια νούμερα. Σύμφωνα με τον είπα το αρμοστή ε, για τους πρόσφυγες. 1.500, μάλλον 15.000, 15.000 άτομα αποβιβάστηκαν. 90% από τις αποβιβάσεις αυτές το 2018 έγιναν στην Τρίπολη. Εμείς 2.000 μπορέσαμε να μετρήσουμε και να τους φροντίσουμε σε, κράτα, κέντρα κράτησης όπου ε, δρούν οι γιατροί χωρίς σύνορα. Ο ίδιος ο ΙΕ τους ε, θεωρεί ότι είναι το 10% περίπου. Δεν υπάρχουν ενελεκτικές επιλογές για τα κέντρα κράτησης. Κάθε προσπάθεια που έγινε, για παράδειγμα, προσπάθεια όπως τελευταία τουλάχιστον για γυναίκες και παιδιά ή πιο, τα πιο ευάλωτα άτομα να μεταφερθούν σε εναλλακτικό ασφαλές κερδοκράτηση. Αυτά απέτυχαν. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Υπάρχει ο ήπατος αρμοστής μπόρεσε ε, να ανοίξει ένα κέντρο που το λέει άφηξη και αναχώρησης. Αυτό συζητήθηκε ως δυνατότητα για κάποια από τα ευάλωτα άτομα που έρχονται από τις αποβιβάσεις για να πάνε στα κέντρα. Αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν τα μοναδικά άτομα που πάνε εκεί είναι αυτά τα οποία έχουν ήδη ενταχθεί σε πρόγραμμα για resettlement. Άλλοι άνθρωποι που έρχονται από τα επιβάσει δεν μπορούν να πάνε στο κέντρο αυτό. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν 70 θέσεις, 70 σε αυτό το κέντρο. Ορισμένες ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις συνεργάζονται με κάποιες υπηρεσίες στέγασης έχουν κάποιες, κάποια, κάποιες δυνατότητες στέγασης δηλαδή, πολύ περιορισμένες, μόνο για γυναίκες με οικογένειες. Αυτό όμως δεν είναι επίσημο πρόγραμμα, δεν αναγνωρίζεται επίσημα δηλαδή. Για αυτά τα άτομα μιλάμε τώρα. 70 θέσεις όλες όλες για εννοητικές δυνατότητες. Προσπαθήσαμε και εμείς να προωθήσουμε λύσεις να πω μονάχα για μια εμπειρία και θα τα πω γρήγορα. Πέρσι τον Ιούνιο διέφυγαν ορισμένοι από, ε, και από σημεία που τους κρατούσαν οι διακινητές και ήρθαν σε εμά. Μπορέσαμε να τους δώσουμε ιατρική βοήθεια. Κάναμε και πιστοποίησαμε κιόλας ότι ήταν θύματα βασανισμών ή πάντως πολύ βαριάς βίαιης ε, ε μεταχείρισης. 50 άτομα ήταν αυτά. Ως γιατροί χωρίς σύνορα, οι ομάδες μας δηλαδή, ήρθαμε σε επαφή με πολλές χώρες για να βρούμε λύσεις για αυτά τα 150 άτομα. Μία ευρωπαϊκή χώρα και μία μη ευρωπαϊκή χώρα δέχτηκαν να βοηθήσουν. Και καμιά από αυτές δεν δέχτηκαν τους ανήλικους. Ενώ μεγάλος αριθμός από τα άτομα αυτά ήταν ανήλικοι. Περάσαμε έξι μήνες για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα άτομα από αυτά, αυτά από τη Λιβύη και είναι ακόμα στον Ήγηρα. Δεν έχουν μπορέσει να ε, μετεγκατασταθούν σε ασφαλή χώρα. Δεν θα πω τώρα στις συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα κράτησης, γιατί νομίζω ότι είναι γνωστές, υπάρχουν πολλές σχετικές εκθέσεις. Αύριο θα δείτε, θα διανύμω έκθεση για την διατροφή σε ένα από τα κέντρα αυτά που νομίζω ότι λέει πολλά από μόνη της. Η δυναμική είναι σημαντική. Ορισμένες από τις συνθήκες έχουν βελτιωθεί κάπως, αλλά η δυναμική παραμένει ίδια. Πριν από λίγες εβδομάδες βρήκαμε άλλο χώρο με 31 άτομα που τα ψάχναμε επί εβδομάδες σε ένα χώρο 4,5 μέτρα επί 5 και χωρίς τουαλέτα, χωρίς τίποτε. Πολύ πρόσφατη εμπειρία αυτή. Το παράδοξο σήμερα ποιο είναι. Το πρόγραμμα IUN έχει καταφέρει να βγάλει ανθρώπους από τη Λιβύη ω εθελοντική επιστροφή. Εμεί το αμφισβητούμε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Μπορέσαμε να του βγάλουμε από τη Λιβύη για αυτούς που δεν θέλουν να μπουν στο πρόγραμμα. Αν είσαστε σε ένα τέτοιο κέντρο και δεν θέλετε να μπείτε, έχετε και του λόγου σα να μην θέλετε να μπείτε στο πρόγραμμα. Όμω άλλη λύση δεν υπάρχει. Είδατε ποιε είναι οι εναλλακτικέ επιλογέ στην κράτηση. Η κατάσταση, τα είπαν και προηγουμένω, είναι ένα σπιράλ ε, ε, επιστροφή στη Λιβύη, επίσημη κράτηση, διαφυγή, διαπόδραση, ε, σύλληψη και ούτω καθεξής. Πολύ περιορισμένες επιλογές λοιπόν που έχουν τα πρόσωπα αυτά. Και κάτι άλλο ακόμη. Το Σεπτέμβριο του 2017 ο ύπατος αρμοστής για τους πρόσφυγες ζήτησε με την κατάσταση 40.000 ατόμων Σεπτέμβριο του 2017 το Γενάρη του 19 εκενώσαμε. Υπάρχει τώρα βέβαια και μια σύγχυση όρων. 40.000 ήταν ο στόχος πάντως. 3.016 άτομα μπόρεσαν να εκενωθούν. Και σε ό,τι αφορά την μετεκατάστασή τους από τη Λιβύη και οι περισσότεροι από αυτούς πήγαν στον Νίγηρα. Μόνο 400 περίπου στην Ιταλία και καμιά κατοστή στη Ρουμανία. και οι τοποθεσίες που έχουν δώσει για αυτό το resettlement, ε, μάλλον οι θέσεις, οι είναι 5.426 ή 56. 5.400 περίπου, επασίλωτος. Αυτή είναι η κατάσταση στη Λιβύη. Ούτε παροχή βοήθειας, ούτε προστασία και πάρα πολύ περιορισμένες οδοί ε, εξόδου, ας πούμε, ή διαφυγής. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Ε, το μόνο που με έρχεται εν πάση στο μυαλό είναι συνενοχή. Σε ένα-δύο λεπτά θα χάσουμε τις διερμηνείς, λέει η Πρόεδρος. Ε, ε, ζητώ συγγνώμη που σας πιέζω, αλλά δεν θα έχουμε άλλη διερμηνία. Κυρία Κατρομπόνη, ευχαριστώ Πρόεδρε. Κατραμπόνε. Οι συνάδελφοι ήδη αναφέρθηκαν στα θέματα που ήθελα και εγώ να αναφέρω και επομένως σε κάποιο βαθμό έχω καλυφθεί. Αλλά ήθελα να αναφερθώ στην ε, παρεμπόδιση των ανθρωπιστικών δράσεων και βοήθεια στην Μεσόγειο. Ελπίζουμε, αν μη τι άλλο, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ξαναεξετάσουν τις δικές τους ευθύνες και τη δική τους αποστολή. Διότι υπάρχει, υφίσταται, παρεμποδίζονται μάλλον οι μη ομίκρον από το να λειτουργούν, να επιχειρούν στη θάλασσα. Αυτό το είπαν όλοι οι συνάδελφοι. Αλλά η δυνατότητα ε, των επιχειρήσεων διάσωσης πρέπει να συνεχιστεί. Το να αφήνουμε απεγνωσμένους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα χωρίς Καμία βοήθεια είναι κάτι το απλά τρομακτικό. Και οι μη σήμερα καλύπτουν ένα κενό. Χρειάζεται λοιπόν μια συντονισμένη στρατηγική για τις επιχείρησεις διάσωσης που θα συμπεριελάμβανε όλες αυτές τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που άκοπα εργάζονται σε αυτό το πεδίο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όμως οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν αποτύχει να σημειώσουν και να αντιμετωπίσουν τα όσα συμβαίνουν στη θάλασσα. Οι διάφορες χώρες δεν έχουν μια συλλογική στρατηγική ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι αρχές του ανθρωπισμού, της ανθρωπιάς, θα γίνονται σεβαστές από όλους. Ποια ήταν η τελευταία φορά που διενήργησαν μια επιχειρήση διάσωσης οι επίσημε αρχέ. Πόσους ανθρώπους έσωσαν το 2018. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση εκατομμυρίων ευρώ καταναλώνεται μόνο, εστιάζεται μόνο στις επιστροφές. Νομίζω ότι τα θεσμικά όργανα που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν τους Ευρωπαίους πολίτες θα πρέπει να αποτυπώνουν ανθρωπιστικές αρχές και να αποτρέψουν τη Μεσόγεια από το να γίνει μαζικός τάφος. Η Ευρώπη μπορεί να σώσει ζωές στη Μεσόγειο και ντούτης δεν έχουμε κανένα συγκεκριμένο project, έργο, για να αναλυφθεί αυτή η ευθύνη. Συζητούμε την μετανάστευση ε, σε ένα πλαίσιο ε, φύλαξης των συνόριων, των συνόρων, ενώ οι ανθρωπιστικές διαστάσεις δεν αναφέρονται ποτέ. Αντί να εστιαστούμε στη διάσωση των ανθρώπων που κινδυνεύουν στη θάλασσα, εστιαζόμαστε στην δημιουργία ενός τείχους, ενός αόρατου τείχους στην Μεσόγειο, που στην ουσία είναι με άλλα λόγια ένα εμπάργκο ναυτικό, θαλάσσιο και το ίδιο εμπάργκο υφίσταται και η δουλειά η δική μας, των ΜΚΟ. Χωρίς να ξεχνούμε την μετεγκατάσταση και την εμπανεγκατάσταση που θα πρέπει να γίνεται με τρόπο οργανωμένο και συντονισμένο. Δεν μπορούμε να αφήνουμε ανθρώπους στο έλεος ε, των κυμάτων ή στο έλεος των σημείων της φύσεως ε, όπως ακούσαμε μαρτυρίες. Η Ευρωπαϊκή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προσφέρει έναν ασφαλή λιμένα. Δεν μπορούμε να αφήνουμε όμως ανθρώπους, γυναίκες και παιδιά στη θάλασσα χωρίς καμία βοήθεια. Άρα το ερώτημά μου και με αυτό κλείνω πρόεδρε είναι τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Λιβύη. Τώρα που η κοινωνία των πολιτών απετράπει από το να διασώζει ανθρώπους που επιχειρούν να διαφύγουν από αυτές τις σκληρές συνθήκες. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιώσει την κατάσταση στη Λιβύη και για να προστατεύσει αθώους που είναι απογεδευμένοι σε αυτή την κόλαση, όπως είπε και η συνάδελφος. Εμείς καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα να επιδείξει μια κάποια ευθύνη και αλληλεγγύη προς τους μετανάστες, προς τους συνανθρώπους μας αυτούς. Η Ευρώπη θα πρέπει να επανέλθει σε επιχειρήσεις διάσωσης, θα πρέπει να καταπολεμήσει τη λαθρεμπορία, των ανθρώπων και θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι διασώσει στη θάλασσα θα διεξάγονται όπως πρέπει να διεξάγονται, χωρίς κενά. Χρειάζεται συνεργασία με τις ΜΚΟ που έχουν αναπτύξει έναν πλούτο εμπειρίας στις θαλάσσιες αυτές επιχειρήσεις διάσωσης και που, έχει δημιουργεί, που έχουν δημιουργήσει μια ζώνη που μπορεί να αντισταθμίσει τις απώλειες ζωής στη θάλασσα. Κανείς που πιστεύει στα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορεί να δεχθεί την εξωτερική ανάθεση, το outsourcing της διαχείρισης των μεταναστών και προσφύγων στη Λιβύη. Πρέπει η νομοθεσία επίσης σχετικά με τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις, τους διαδρόμους τους ανθρωπιστικούς να επικαιροποιηθούν. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτήν την τρομακτική οδύσσια που περνούν οι άνθρωποι αυτοί για να βρουν ένα, έναν ασφαλή λιμένα, ένα καλύτερο μέλλον. Το πολιτικό συμφέρον δεν θα πρέπει να προηγείται των ανθρώπων και, των, και της ζωής τους. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ε, πολύ λυπούμε που έχουμε πλέον αφόρητη πίεση χρόνου. συνάδελφοι, εφτάσαμε στο τέλος αυτής της δεύτερης συνεδρίασης. Έχουμε ήδη υπερβεί το χρονοδιάγραμμα δεν πρόκειται να προβώ σε κανένα συμπέρασμα αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές, ε, τον Dietmar Κώστερ, ε, από το απόγευμα όλους τους προηγούμενους ομιλητές, εκπροσώπους των ΜΚΟ, όλους τους συναδέλφους που παρενέβησαν. Δεν θα δώσω εγώ κάποιο συμπέρασμα ακούσαμε τις μαρτυρίες των εκπροσώπων των ΜΚΟ και αυτές οι μαρτυρίες μιλούν από μόνες τους. Και ο Φιλίμων Μομπρετών μας έδωσε μια μαρτυρία που πραγματικά πρέπει να είναι κατανοητή για όλους. Όταν μας είπε ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει την αξιοπρέπεια να αναγνωρίζεται ως ίσος με τους άλλους. Ως μετανάστης και εγώ Αντιλαμβάνομαι τι λέει. Ο ρατσισμός είναι μια λέξη που δεν ακούστηκε καθόλου σήμερα, αλλά είναι ένα φαινόμενο στην καρδιά του, φαινο, του της προσέγγισής μας προς τους ανθρώπους αυτούς. Τους βλέπουμε ως κάτι διαφορετικό. Αν τους βλέπαμε ως ίδιους με μας δεν θα πέθαιναν σε τόσο μεγάλους αριθμούς και το λέω με σαφήνεια. Αυτό βρίσκεται πίσω από τα κρούσματα αυτά η Κάθριν Σμιτ είχε δίκιο όταν είπε ότι είναι ηρωνικό που έρχεται στο κοινοβούλιο για να μας ε, ε, δώσει σκληρά διδάγματα. Αλλά στην πραγματικότητα στο κοινοβούλιο βλέπουμε πολλές φωνές φιλελεύθερες, πολλές φωνές ανθρώπων που υποπίεση προσπαθούν να κάνουν αυτό που πρέπει. Είναι σημαντικό λοιπόν τα μηνύματα αυτά να ακούγονται εδώ μέσα να ακούγονται οι μαρτυρίε των ανθρώπων που έχουν δραστηριοποιηθεί στο πεδίο. Θα δώσω απλώς ένα παράδειγμα, την ε, δίωξη της ε, παροχής βοήθειας συνδρομής ανθρωπιστικής. Προσπαθούμε να οθήσουμε το Κοινοβούλιο προ την κατεύθυνση αυτή. Σε αυτό το σημείο δυστυχώς η διερμηνία τερματίζεται. Καλό σας βράδυ